εγκρίνονται. Ανακοινώσει του Πρόεδρου. Η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά και η Σκανδιναβική Αριστερά έχουν έρθει σε επαφή με το Προεδρείο για τον ορισμό κάποιων μελών και αν δεν υπάρχει κάποια παρατήρηση ή ένσταση τότε ε,